Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε. Όπως γνωρίζετε, σήμερα η μερίσια διάταξη προβλέπει την δήλωση της προταθήσης υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι για αυτή τη διαδικασία δεν προβλέπεται το περίφημο Catch the Eye, ούτε η επίδειξη των μπλε καρτών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φόντερ Λάιεν για να ακούσουμε τη δήλωσή της. Πριν από ακριβώς 40 χρόνια, η πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Σιμών Βέιλ, εξελέγει και παρουσίασε το δικό της όραμα για μια Ευρώπη πιο ενωμένη και πιο δίκαιη. Χάρη σε αυτήν και χάρη σε όλες τις άλλες εμβληματικές ευρωπαϊκές φυσιογνωμίες, σήμερα σας παρουσιάζω το όραμα που έχω εγώ για την Ευρώπη. Και 40 χρόνια αργότερα, με μεγάλη περηφάνεια μπορώ να πω, επιτέλους μία γυναίκα θα είναι υποψήφια για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι υποψήφια χάρη σε όλους αυτούς και όλες εκείνες που κατέριψαν φραγμούς και συμβάσεις. Είμαι υποψηφία χάρη σε όλους αυτούς και όλες εκείνες που οικοδόμησαν μια Ευρώπη ειρήνης, μια Ευρώπη ενωμένη και μια Ευρώπη αξιών αυτή η ευρωπαϊκή ε, πεποίθηση με ε, καθοδήγησε σε ολόκληρη τη ζωή μου και στην καριέρα μου ως μητέρα, ως γιατρό αλλά και ως ε, γυναίκα πολιτικό. Και αυτό το θάρρος, αυτή η τόλμη των πρωτοπόρων όπως η Σιμών Βέιλ βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο του οράματος που έχω για την Ευρώπη. Και αυτό το πνεύμα θα καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας έχω την πρόθεση να προεδρεύσω. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι πατέρες και οι μητέρες της Ευρώπης από τη στάχτη και τα ερήπια των παγκοσμίων πολέμων κατόρθωσαν να επιτύχουν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και αυτό είναι η ειρήνη μια κοινή αγορά, εμπόριο χωρίς φραγμούς, ταξίδια, έρευνα, εργασία. Έχουμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους οι οποίοι σήμερα ζουν από τη Ρήγα μέχρι τη Λεμεσό, από την Αθήνα μέχρι τη Λισαβόνα και όλοι ζουν ε, με ειρήνη και ευημερία. Η γενιά των δικών μου των παιδιών ε, δεν μπορεί να φανταστεί ε, μια Ευρώπη χωρίς αυτό το αίσθημα της πατρίδας. Όταν λοιπόν γεννήθηκε αυτή η ευτυχισμένη γενιά και εμείς οι πιο ηλικιωμένοι είχαμε σκεφτεί ότι τα πράγματα θα ακολουθήσουν αυτή την πεπατημένη. Σήμερα όμως όλοι πια γνωρίζουν ότι πρέπει να ξανά αγωνιστούμε, να αντισταθούμε για την Ευρώπη μας ε, Στον κόσμο ολόκληρο βλέπουμε καταστροφικές εξελίξεις οι οποίες δεν μπορούν να αφήσουν ανέγκυχτη την Ευρώπη. Βιώνουμε τη δημογραφική αλληλήγη αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση, την ταχύτατη ψηφιοποίηση του κόσμου της εργασίας και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Καμία από αυτές τις μεταεξελίξεις δεν είναι καινούρια. Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν προβλεφθεί εδώ και καιρό από την επιστήμη. Εκείνο όμως που είναι καινούριο είναι ότι σήμερα ως πολίτες Ευρώπης, ανεξάρτητα με το σε ποια χώρα ζούμε, βιώνουμε στο πετσί μας τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων. Είτε πρόκειται Πρόκειται για τους Φινλανδούς αγρότες ε, σιτηρών και καλλιεργητές ε, αγροτικών προϊόντων που ε, παιδεύονται, τυρανιώνται από την ξηρασία έως και πολλές άλλες εξελίξεις. Όλα τα βιώνουμε όπως σας είπα στο πετσί μας. Όμως πρέπει να γνωρίζουν όλοι και οι συνταξιούχοι στην Ιρλανδία αλλά και όσοι θέλουν να έχουν απευθείας και ηλεκτρονικές τραπεζικές συλλαγές, συναλλαγές ότι πρέπει να εξοικειωθούν με αυτές τις εξελίξεις. Είτε πρόκειται για νοσοκομεία που πρέπει να κλείσουν είτε για άλλες δημογραφικές εξελίξεις όλοι το βιώνουμε στις δικές μας εμπειρίες και όλα αυτά άφησαν τους ανθρώπους με την αίσθηση ότι χάνουν τον έλεγχο. Καμιά από αυτές τις προκλήσεις δεν θα απομακρυνθεί αλλά είχαμε διαφορετικούς τρόπους να αντιδράσουμε σε αυτές τις τάσεις. Κάποιοι στρέφονται προς αυταρχικά καθεστώτα, άλλοι αγοράζουν την παγκόσμια επιρροή τους και δημιουργούν εξαρτήσεις, επενδύοντας σε λιμάνια και δρόμους και άλλοι στρέφονται προς τον προστατευτισμό. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν είναι για μας. Εμείς θέλουμε πολυμέρεια, θέλουμε δίκαιο εμπόριο. Είμαστε υπέρ της τάξης με βάση τους κανόνες, διότι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι καλύτερο για όλους μας. Θα πρέπει να το κάνουμε με τον ευρωπαϊκό τρόπο. Αλλά αν θα ακολουθήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό μονοπάτι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξαναανακαλύψουμε τη δική μας ενότητα. Εάν είμαστε ενωμένοι από μέσα, κανείς δεν θα μπορεί να μας χωρίσει απ' έξω. Εάν κλείσουμε τα χάσματα ανάμεσά μας, θα, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις του σήμερα στις ευκαιρίες του αύριο. Αξιότιμα μέλη η πιο ισχυρή μας πρόκληση είναι να διατηρήσουμε την υγεία στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη και ευκαιρία των καιρών μας. Θέλω η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη ήπειρος ε, ουδέτερη από πλευράς κλίματος μέχρι το 2050. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τολμηρά βήματα όλοι μαζί. Ο στόχος που έχουμε σήμερα για τη μείωση των εκπομπών κατά 40% μέχρι το 2030 δεν επαρκεί. Θα πρέπει να πάμε παραπέρα, θα πρέπει να αγωνιστούμε για περισσότερο. Μία προσέγγιση σε δύο βήματα απαιτείται για να μειώσουμε τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 κατά 50, εάν όχι και 55%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ηγείται των διεθνών διαπραγματεύσεων για να αυξήσει το επίπεδο φιλοδοξίας άλλων μείζων οικονοποιών μέχρι το 2021. Γιατί για να πετύχουμε πραγματικό αντίκτυπο δεν πρέπει απλά να είμαστε φιλόδοξοι εδώ στο σπίτι μας. Ναι, θα πρέπει να το κάνουμε, αλλά πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί. Και για να το πετύχουμε αυτό, θα προτείνω μία πράσινη συμφωνία για την Ευρώπη στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας μου. Θα προτείνω την το πρώτο νόμο περί κλίματος στην Ευρώπη που θα θέσει τον στόχο του 2050 σε νόμο. Αυτή η αύξηση της φιλοδοξίας θα χρειαστεί επένδυση, ε, μίζωνα επένδυση. Τα δημόσια κονδύλια δεν θα επαρκούν. Θα προτείνω ε, ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο και θα μετατρέψω ε, μέρη της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας σε μια τράπεζα του κλίματος. Αυτό θα ξεκλειδώσει ένα τρισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεων για την επόμενη δεκαετία. Αυτό σημαίνει αλλαγή. Όλοι μας και κάθε τομέα θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό. Από την αεροπορία μέχρι τις θαλάσσιες μεταφορές, μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας ταξιδεύει και ζει. Οι εκπομπές θα πρέπει να έχουν μια τιμή που να αλλάξει την ε, συμπεριφορά μας. Και για να συμπληρώσω αυτό το έργο και για να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε μας μπορούν να συναγωνίζονται επίσης όρις, θα εισαγάγω έναν συνοριακό φόρο του άνθρακα για να αποφεύγονται οι διαρροές άνθρακα. Αξιότιμα μέλη, αυτό που είναι καλό για τον πλανήτη μας θα πρέπει να είναι καλό και για τους ανθρώπους και για τις περιφέρειές μας. Ασφαλέστατα και γνωρίζω την σημασία των ταμείων συνοχής. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη μετάβαση για όλους. Δεν έχουν όλες οι περιφέρειες την ίδια αφετηρία. αλλά όλοι έχουμε τον ίδιο προορισμό. Είναι γι' αυτό που προτείνω ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης για να στηρίξω αυτούς που επηρεάζουν περισσότερο. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκό τρόπο. Είμαστε φιλόδοξοι και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω και προσφέρουμε προοπτικές. Εάν θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, χρειαζόμαστε μια ισχυρή οικονομία. Γιατί αυτό που θέλουμε να δαπανίσουμε πρέπει πρώτα απ' όλα να το κερδίσουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι καινοτόμε, είναι επιχειρηματικές, είναι ευέλικτες, ευκάμπτες, δημιουργούν θέσεις επασχόλησης, παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στους νέους μας αλλά μπορούν να το κάνουν αυτό μόνο εάν έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια παντού σε αυτή την τεράστια νέα αγορά. Ας απαλλαχτούμε από τους φραγμούς, ας ανοίξουμε την πόρτα, ας ολοκληρώσουμε επιτέλους την ένωση των κεφαλαίων αγορών, γιατί το αξίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Και πρέπει να δουλέψουμε εντός του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εκεί που χρειάζονται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη την ευελιξία που επιτρέπουν οι κανόνες. Είμαστε περήφανοι για τις οικονομίες μας, θέλουμε να τις ενισχύσουμε. Αλλά υπάρχει και μια σαφής λογική. Δεν είναι οι άνθρωποι που εξυπηρετούν την οικονομία μας, είναι η οικονομία που εξυπηρετεί τους ανθρώπους μας. Στην ε, η οικονομία της, κοινων... αγοράς θα πρέπει να συμφιλιώσουμε την αγορά με το κοινωνικό. Άρα θα επαναστιάσω το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο για να διασφαλίσω ότι ακολουθούμε τους στόχους αηφόρους ανάπτυξης και θα είμαι υπέρ δίκαιων φόρων. Είτε μιλάμε για τις οικοδομές ή για τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Όταν οι γίγαντες της τεχνολογίας κάνουν τεράστια κέρδη στην Ευρώπη, αυτό είναι πολύ καλό γιατί είμαστε μια ανοιχτή αγορά και μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά εάν κάνουν αυτά τα κέρδη ε, εποφελούμενοι των εκπαιδευτικών συστημάτων μας, των ε, εργαζομένων μας, των υποδομών μας και της κοινωνικής ασφάλισης, αν αυτό ισχύει, τότε δεν είναι αποδεκτό να κάνουν αυτά τα κέρδα και, κέρδη και να μην πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους, γιατί παίζουν με το φορολογικό μας σύστημα. Αν θέλουν να υποφαληθούν, θα πρέπει να μοιραστούν και το βάρος. Αξιότιμα μέλη, ο ευρωπαϊκός τρόπος αφορά προφανώς και το να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο του δυναμικού μας. Το δυναμικό μας είναι οι άνθρωποι, οι δεξιότητές μας, ε, η διαφορετικότητα που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε στο να έχουμε μια πιο δίκαιη, πιο ισότιμη Ευρώπη και αυτό θα είναι το κίνητρό μου κάθε μέρα που θα είμαι στο αξίωμά μου. Όπω συνέβη και καθ' όλη τη διάρκεια τη σταδιοδρομία μου. Έχω διανύσει μια μακρά πορεία. Ήμουν υπουργό οικογένεια και αγωνίστηκα για να μπορέσω να θεσπίσω τι ε, γονεϊκέ άδειε. Όμω ο αγώνα για τη δικαιοσύνη ποτέ δεν σταματά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για οικογένειε που δουλεύουν σκληρά. Είναι ακόμα δύσκολο να τα καταφέρουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να διασφαλίσω ότι η εργασία θα αμείβεται σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς κάθε άνθρωπος που δουλεύει με πλήρη απασχόληση θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει ένα κατώτατο εισόδημα για να βιοπορίζεται με αξιοπρέπεια. Ως εκ τούτου θα αναπτύξουμε ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο που βέβαια θα σέβεται τις διαφορετικές αγορές εργασίας. Αλλά πιστεύω ότι η βέλτιστη λύση είναι να έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις όπου θα συμμετέχουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι γιατί αυτό ...τι θα προσαρμόσουν τον κατώτατο μισθό ανάλογα με την περιοχή. Βεβαίω και γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα, αλλά εμεί πρέπει να καθορίσουμε το πλαίσιο. Και επιθυμώ μια καλύτερη προστασία για εκείνου που χάνουν τη δουλειά του οποτεδήποτε πλήτεται η δική μα οικονομία. Ευρωπαϊκό σύστημα εξασφάλιση επιδομάτων ανεργία. Θα στηρίξουμε του ανθρώπου μα οποτεδήποτε προκύπτουν εξωτερικά οικονομικά σοκ. Βεβαίω και υπάρχουν εθνικά εθνικά συστήματα ασφάλισης. Όμως αυτό το σύστημα της εξασφάλισης, της αντασφάλισης αν θέλετε, είναι ένα σύστημα που είναι επιγόντως απαραίτητο στην Ευρώπη. Επιθυμώ επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα και δικαιοσύνη για τους νέους ανθρώπους. Ε, περίπου 14% οι μάλλον για να το πω αλλιώ, η ενεργία των νέων κυμαίνεται από 5 μέχρι 40% σε κάποιε χώρε. Οι νέοι όμω έχουν φιλοδοξίε. Θέλουν να δουλέψουν, να έχουν εξασφαλισμένο μέλλον. Δική μα είναι η δουλειά να του βοηθήσουμε να το επιτύχουν. Και γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω την, ε, το εργαλείο εγγύηση για του νέου. Αυτό το είχα πρωτοεμφανίσει στη Γερμανία όταν ήμουν αρμόδια υπουργό και νομίζω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα στηρίξω αυτά που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο προπολογισμό για το πρόγραμμα Εράσμους να τριπλασιαστεί κατά την επόμενη περίοδο όταν θα σχεδιαστεί ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε να μεριμνούμε για τους πλέον ευάλωτους, που είναι τα παιδιά μας. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Το γνωρίζω. Είμαι μητέρα 7 παιδιών και ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά το να μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στη μουσική, σε υγιεινή διατροφή και σε ένα καλό περιβάλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν το εργαλείο εγγύηση για τα παιδιά έτσι ώστε κάθε παιδί στην Ευρώπη να είναι προστατευμένο από τη φτώχεια και από τον κοινωνικό ε, αποκλεισμό. Να έχει δικαίωμα στην παιδεία και την υγεία. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ θα και θα φροντίσω να εξασφαλιστούν όλα αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του προγράμματός μου ε, να ε, δώσω ζωή στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θα ξεκινήσω δίδοντας βέβαια το καλό παράδειγμα ε, και θέλω να πω τι σημαίνει, σημαίνει ότι στο Κολέγιο των Επιτρόπων θα εξασφαλίσω ώστε να υπάρχει πλήρης ισότητα των δύο φύλων. Εάν τα κράτη-μέλη δεν προτείνουν αρκετές γυναίκες επιτρόπους, δεν θα διστάσω να ζητήσω νέα ονόματα, νέους υποψηφίους. Από το 1958 είχαμε 183 επιτρόπους και μόνο 35 εξ αυτών ήταν γυναίκες, δηλαδή λιγότερο από το 20% αλλά εμείς εκπροσωπούμε το ίμιση του πληθυσμού. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε αυτό που μας αξίζει. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για τη βία κατά των γυναικών. Εάν μία στις πέντε γυναίκες έχει ήδη υποστεί ε, σεξουαλική και σωματική βία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το 55% των γυναικών υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση, προφανώς αυτό δεν είναι μόνο θέμα γυναικών. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα προτείνω η βία κατά των γυναικών να προσθεθεί στον κατάλογο των ε, εγκλημάτων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της ανθρωπότητας και να προσθεθεί το θέμα αυτό στη συνθήκη. Είμαι πεπισμένη ότι αν μπορέσουμε να κλείσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ημών, τότε θα ανακύψουμε, θα εμφανιστούμε ως μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Αξιότιμα μέλη. Η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η ελληνική φιλοσοφία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Και η ευρωπαϊκή μας ε, Ήπειρος ε, πέρασε ε, σκοτεινές περιόδους όταν την εξουσία την είχαν δικτάτορες και όταν είχε καταργηθεί το κράτος δικαίου. Για πάρα πολλούς αιώνες οι Ευρωπαίοι αγωνίστηκαν σκληρά για την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία τους. Το κράτος δικαίου είναι το καλύτερο εργαλείο για να προστατεύσουμε τις ελευθερίες μας και να προστατεύσουμε κυρίως τους ευάλωτους στην Ευρώπη. Και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί θέμα συμβασμού. Δεν υπάρχει θέμα συμβασμού όταν το διακύβευμα είναι το κράτος δικαίου. Και δεν θα υπάρξει ποτέ. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλη την εργαλειοθήκη που διαθέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτύχουμε το στόχο μας. Εγώ θα στηρίξω έναν ενωσιακό μηχανισμό κράτους δικαίου. Και για να είμαι απόλυτα σαφή ε, το νέο αυτό εργαλείο δεν είναι εναλλακτική λύση αυτά που ήδη υπάρχουν, απλά είναι μία προσθήκη στα ήδη υπάρχοντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θα είναι ανεξάρτητος θεματοφύλακας ε, των συνθήκων. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή και η δικαιοσύνη θα υπερασπίζεται το κράτος δικαίου οπουδήποτε και οποτεδήποτε αυτό υφίσταται επιθέσεις. Αξιωτούμε μέλη, το κράτος δικαίου είναι κάτι το καθολικό που εφαρμόζεται σε όλους. Τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 17.000 άτομα πνίγηκαν στην Μεσόγειο. Η Μεσόγειος έχει καταστεί ένα από τα πιο θανάσιμα σύνορα στον κόσμο. Στη θάλασσα υπάρχει το καθήκον διάσωσης των ζώων, αλλά και στις ε, συμβάσεις μας υπάρχει το νομικό και ηθικό καθήκον για τον σεβασμό της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπινου όντως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να προασπίζεται αυτές τις αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σύνορα με ανθρώπινο πρόσωπο. Θα πρέπει να διασώζουμε ε, αλλά η διάσωση δεν αρκεί. Θα πρέπει να μειώσουμε την παράτυπη μετανάστευση, να καταπολεμήσουμε τους λαθρεμπόρους και τους διακινητές, το οργανωμένο έγκλημα, να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στο άσυλο, να βελτιώσουμε την κατάσταση των προσφύγων. Για παράδειγμα, με ανθρωπιστικούς διάβλους σε συνεργασία με το UNHCR. Χρειάζεται να έχουμε ενσυναίσθηση και αποφασιστική δράση. Γνωρίζω πόσο δύσκολες και πόσο διχαστικές είναι οι συζητήσεις στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις νόμιμες ανησυχίες των πολλών και να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Εγώ θα προτείνω ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που να περιλαμβάνει και την επανεκκίνηση της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου. Αυτό θα μας επιτρέψει να επανέλθουμε σε μια πλήρως ε, λειτουργική, ε, ένα, χώρο Σέγγεν πλήρω λειτουργικό με ελευθερία κίνησης, το, κλειδί στην ευημερία μας, στην ασφάλεια και τις ελευθερίες. Ε, υπάρχει ε, στο κέντρο αυτό η επανενίσχυση της Ευρωπαϊκής Σύνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σώμα των 10.000 ε, σύνοριοφυλάκων της του Frontex μέχρι το 2024 σίγουρα. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε το σύστημα ασύλου μας. Ένα κοινό σύστημα ασύλου θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να πετύχουμε, να είναι κοινό. Μπορούμε να έχουμε σταθερά εξωτερικά σύνορα μόνο εάν δώσουμε αρκετή βοήθεια στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση για, ε, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Χρειάζεται αλληλεγγύη. Πρέπει να αλληλοβοηθηθούμε και να συνεισφέρουμε. Χρειάζεται ένας νέος τρόπος επιμερισμού του βάρους και θα πρέπει να κάνουμε δίκαιες προσφορές συνεργασίες σε χώρες προέλευσης και μετάβασης που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Διπλωματία, οικονομική ανάπτυξη, επένδυση, σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά απαιτούνται έτσι ώστε να έχουν κάποια προοπτική οι άνθρωποι. Θα ήθελα να σας πω μια ιστορία για αυτό το θέμα της προοπτικής. Πριν από τέσσερα χρόνια Ήμουν τυχερή γιατί ε, φιλοξενήσα ένα 19χρονο πρόσφυγα από την Συρία στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Δεν μιλούσε καθόλου γερμανικά και ήταν ε, βαθιά πληγωμένος από την εμπειρία του εμφυλίου πολέμου στη χώρα του και της φυγής, της προσφυγοποίησης του. Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια, μιλάει άπτεστα γερμανικά, αγγλικά, φυσικά μιλάει και τα αραβικά είναι ε, την ημέρα ε, για τις, ε, στην κοινότητά του και κάνει επαγγελματική κατάρτιση και παρακολουθεί και μαθήματα δευτερομάθημιας εκπαίδευσης το βράδυ. Είναι μια έμπνευση για όλους μας και μια μέρα θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του. Αξιότιμα μέλη, ως Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκα πολλές φορές αυτή την εμπόλεμη γειτονία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του πρώην Προέδρου του Ιράκ, του Μασούμ, που είχε πει «Θέλουμε να δούμε περισσότερη Ευρώπη εδώ πέρα». Ο κόσμος καλεί για περισσότερη Ευρώπη, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη φωνή στον κόσμο και χρειάζεται να δράσει γρήγορα. Γι' αυτό είναι που πρέπει να έχουμε το κουράγιο να πάρουμε αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής με πλειοψηφία και να σταθούμε ενωμένοι σε αυτές τις αποφάσεις μας. με ενισχυμένη πλειοψηφία πρέπει να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συλλογική άμυνας μας θα είναι πάντα το ΝΑΤΟ. Θα παραμείνουμε διατλαντικοί, αλλά και πρέπει να είμαστε, καταστούμε όμως πιο Ευρωπαίοι. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση Άμυνας. το έργο μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας ενσωματώνεται σε μια συνολική ασφάλεια. Η σταθερότητα, η αστεθεροποίηση πάντα συνοδεύεται με την διπλωματία, την επανασυμφιλίωση και την ανοικοδόμηση οι άνδρες και οι γυναίκες μας των ενόπλων δυνάμεων δουλεύουν δίπλα στους αστυνομικούς, στους διπλωμάτες και τους εργαζόμενους στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και αξιότιμα μέλη, αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες αξίζουν τον πλήρη σεβασμό μας και την αναγνώρισή μας για τις ε, αδιάκοπες ε, προσπάθειες που κάνουν για προς την Ευρώπη. Δεν μπορώ να μιλήσω για την Ευρώπη χωράς να μιλήσω και για τους φίλους μας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για πρώτη φορά το 2016 ένα κράτος μέλος αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. This is... Πρόκειται για μια σοβαρή απόφαση. Λυπούμαστε γι' αυτό αλλά σεβόμαστε αυτή την απόφαση. Από τότε, μαζί με την τρέχουσα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να ε, διοργανώσει την ομαλή, την εύκτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία αποχώρησης που συνάφθηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ε, ε, σιγουριά εκεί όπου το Brexit δημιούργησε ανασφάλεια, διατηρώντας ε, τα δικαιώματα των πολιτών και διατηρώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί της Ιρλανδίας. Αυτές οι δύο προτεραιότητες είναι και δικές μου προτεραιότητες. Ωστόσο, είμαι έτοιμη για περαιτέρω παράταση της ημερομηνία απαχώρησης εάν χρειαστεί και απαιτείται περισσότερος χρόνος για, ένα, για κάποιο καλό λόγο. In Εν πάση περιπτώσει, σε οποιαδήποτε περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει σύμμαχός μας, εταίρος μας ε, και φίλος μας. Αξιότιμα μέλη, όταν ε, ήρθα στο Στρασβούργο πριν από 13 ημέρες υποσχέθηκα ότι ήρθα για να ακούσω. Άκουσα τις ανησυχίες σας, ε, τις ε, ελπίδες σας, ε, τις προσδοκίες σας, οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που σας έστειλα αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις μας. Και από όλα αυτά που άκουσα κατέληξα σε συμπεράσματα και έλαβα τις αποφάσεις μου. Πρώτα απ' όλα, επιθυμώ οι Ευρωπαίοι πολίτες να διαδραματίσουν καθοριστικό και ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ένωσης μας, της Ευρώπης μας. Θέλω οι πολίτε ε, να έχουν λέγει σε μια συνδιάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη ε, που θα ήθελα να ξεκινήσει το 2020 και να διαρκέσει δύο χρόνια. Δεύτερον, επιθυμώ να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα των Spitzenkandidaten, των κορυφαίων υποψηφίων. Αυτό το σύστημα πρέπει να είναι περισσότερο ορατό σε ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των υπερεθνικών εκλογικών καταλόγων ε, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκλογών, έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και τρίτον, ναι, πράγματι υποστηρίζω το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν το σώμα αυτό με την δική του την πλειοψηφία υιοθετεί ψηφίσματα που καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα ακολουθούν νομοθετικές πράξεις που θα σέβονται την αναλογικότητα, την επικουρικότητα και την αρχή της καλύτερης νομοθεσίας. Είμαι πεπισμένη ότι η σχέση μας, η ισχυρότερη σχέση μας με τους εταίρους μας θα βοηθήσει έτσι ώστε να ακούγεται καλύτερη φωνή μας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ο πατέρας μου ήταν 15 ετών όταν ο Φρικαλαίος πόλεμος που επέφερε στην ε, στην Ήπειρό μας το θάνατο, τον όλεθρο, την προσφυγιά όταν τέλειωσε αυτός ο πόλεμος. Ο πατέρας μου λοιπόν ε, πολλές φορές αναφερόταν σε αυτόν τον πόλεμο, σε μένα και στα υπόλοιπα έξι παιδιά του και πολύ συχνά μας έλεγε το τι σήμαινε για εκείνον το γεγονός ότι άλλες χώρες ε, βοήθησαν, μας έτειναν χείρα βοηθείας για να μας συμπεριλάβουν στον κύκλο των δημοκρατικών κρατών. Ο πατέρας μου άρχισε να εργάζεται στην ΕΚΑΧ, την Ένωση, την Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Είπε τότε ότι επιτέλους αρχίζει το εμπόριο και όταν υπάρχουν εμπορικές ανταλλαγές, τότε οι διαπραγματευόμενοι αναπτύσσουν ε, φιλικές σχέσεις και δεν καταπολεμούν και δεν σκοτώνουν ένα τον άλλο. Ο πατέρας μου ήταν στην αρχή διευθυντής του γραφείου Γερμανού Διπλάτη διπλωμάτη του Φόντερ Γκρόμπεν και αργότερα έγινε γενικό διευθυντή στην Γενική Διεύθυνση Θεμάτων Ανταγωνισμού. Εγώ γεννήθηκα εδώ στι Βρυξέλλες και γι' αυτό είμαι Ευρωπαία και αργότερα έμαθα ότι είμαι Γερμανίδα και κατάγομαι από την κάτω Σαξονία. Για μένα υπάρχει ένα μόνο πράγμα. Πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη. Όποιο λοιπόν θέλει μαζί μου να βοηθήσει στο να ενισχυθεί η Ευρώπη, όλοι αυτοί θα με έχουν στο πλευρό τους ως παθιασμένη αγωνίστρια. Όποιος όμως θέλει να αφαιρέσει από την Ευρώπη τις αξίες της ε, θα βρει στο πρόσωπό μου μία ορκισμένη εχθρό. Όταν ο πατέρας μου πλέον ε, ήταν πολύ ηλικιωμένος ε, και έφτανε στο, στη δύση της ζωής του, τότε άλλαξε και το αφήγημά του για την Ευρώπη. Ο πατέρας μου τότε δεν μιλούσε πια τόσο πολύ για τον πόλεμο, τότε πια έλεγε ότι η Ευρώπη είναι όπως ένας μακροχρόνιος γάμος. Δηλαδή η αγάπη δεν αυξάνεται όλο και περισσότερο, δεν είναι όπως την πρώτη μέρα, όμως η αγάπη γίνεται πιο βαθιά. Πιο βαθιά και ξέρει κανείς ότι μπορεί να βασιστεί στον άλλον σε καλούς και σε χαλεπούς καιρούς. Γνωρίζει κανείς ότι μπορεί να τσακώνεται, αλλά θα τα ξαναβρει, θα συμφιλειωθεί και ποτέ δεν ξεχνά κανείς γιατί α, θελήσαμε αυτό το δεσμό. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ σε αυτήν την αίθουσα ζούμε σε μια Ευρώπη που έγινε πιο όρημη, που μεγάλωσε, που είναι πολύ ισχυρή με 500 εκατομμύρια κατοίκους ε, πάνω από 200 εκατομμύρια προσήλθαν στι κάλπε. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη έχει επιρροή. Αυτή η Ευρώπη θέλει να αναλάβει ευθύνη. Ευθύνη για την ίδια και για τον κόσμο. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Το γνωρίζω πολύ καλά. Πονάει. Είναι δύσκολο. Όμω αυτό είναι το πιο ευγενικό καθήκον μα. Οι νέοι θέλουν να προχωρήσουν. Τα δικά μου τα παιδιά μου λένε και δικαίω, μα μην περιμένετε να περάσει απλά ο καιρό. Κάντε κάτι και γι' αυτό το λόγο εγώ έθεσα υποψηφιότητα. Γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σα και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο καλώ όλους τους Ευρωπαίους να με στηρίξουν γιατί είναι το πιο πολύτιμο αυτό που έχουμε. Ζήτω η Ευρώπη, Bible Hope, Long Live Europe. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie. Ευχαριστώ πολύ την κυρία der Leyen για την εισήγησή της. Ε, τώρα θα δώσουμε τον λόγο στους προέδρους ε, των ε, πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσω με τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Μάνφρεντ, έχεις τον λόγο. Αξιότιμη κυρία Φόντα Λάιεν, αξιότιμη πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Μετά την εκλογή του πρόεδρου μας πριν από δύο εβδομάδες, τώρα έχουμε μπροστά μας την εκλογή Τη Προέδρου τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την κυρία Φοντελάιν για το πρόγραμμα που παρουσίασε, για τι προτάσει της για το μέλλον τη Ευρώπη. Για μας, ε, την πολιτική μα ομάδα του ΕΛΚ, ε, αυτό που έχει σημασία είναι οι υποσχέσεις που δώσαμε στου πολίτε. Οι πολίτες, οι υποσχέσεις αυτές είναι για μα το σημείο προσανατολισμού. 40 εκατομμύρια πολίτε ψήφισαν τους δικού μα τους ευρωβουλευτέ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Αυτοί λοιπόν περιμένουν από εμάς τα θέματα τα οποία τους τα υποσχεθήκαμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Μια δίκαιη Ευρώπη όπου οι συνθήκες διαβίωσης θα μοιάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια σύγχρονη Ευρώπη όπου ε, θα προωθηθεί, θα ενισχυθεί η έρευνα. Μια ασφαλή Ευρώπη όπου τα σύνορα θα είναι πιο ασφαλή κατά της παράτυπης ε, μετανάστευσης. Μια ανοιχτή Ευρώπη που θα κάνει εμπορικές ανταλλαγές, θα έχει σχέση με την Αφρική και μια οικολογική Ευρώπη που θα προστατεύει το κλίμα μας και που ε, θα έχει πάντα κατά νου τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Η Ursula von der Leyen είναι χριστιανοδημοκράτης, είναι πεπισμένη φιλοευρωπαία και γι' αυτό από κοινού θα εφαρμόσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σήμερα θα ψηφίσει για την Ursula von der Leyen στο σύνολό του και θα ήθελα να απευθυνθώ στην Σκακέλερ και σε άλλους. Για αυτά τα έχουν προτείνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η άμυλα ε, του να είναι κανείς ε, υποψήφιος, ε, να προσπαθήσει να αγωνιστεί για τις απόψεις του, να προσπαθήσει να πείσει ανθρώπους και μετά ως δημοκράτης να σέβεται το αποτέλεσμα. 201 εκατομμύρια άνθρωποι όπως σας είπα, προσήλθαν στις κάλπες τις ευρωπαϊκές εκλογές. Μα ποιο, πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εορτή. Και όλοι αυτοί θέλουν μια δημοκρατική Ευρώπη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών κατέδειξαν με απόλυτη σαφήνεια ότι δυστυχώς πολλές φορές αγνοείται η θέληση των ανθρώπων. Γιατί είχαμε, παραδείγματος χάνει δημοκρατικά προτινόμενους υποψήφιους, οι οποίοι για καθαρά κομματικούς λόγους χαρακτηρίστηκαν ε, ως μη εκλόγιμοι. Ε, αυτό ήταν ζημιά για τη δημοκρατία. Και τη ζημιά αυτή δεν μπορεί κανεί να την επουλώσει προκαλώντας νέε ζημιέ. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα την πράξη, χρειάζεται σταθερότητα. Γι' αυτό το λόγο η δική μου πολιτική ομάδα πριν από δύο εβδομάδες ε, ε, στήριξε ε, τον κύριο Σασόλη, τον υποψήφιο των Σοσιαλδημοκρατών και σήμερα περιμένω ως πρόεδρος του ΕΛΚ και η άλλη πλευρά να στηρίξει την κυρία Ούρσουλα Φόντελάν στη θέση της υποψηφίου του, ε, του, του υποψηφίου πρόεδρου. Και σας λέω, μόνο αν ο ένας στηρίζει τον άλλο, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Βεβαίως, τα επόμενα πέντε έτη πρέπει να λειτουργήσουμε ε, με την έννοια της Δημοκρατικής Ευρώπης, να έχουμε νομοθετικές δυνατότητες και πρωτοβουλίες, να εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο και να υπάρχει και η νομική κατοχήρωση Τη ε, πρόταση του Spitzenkandidat έτσι ώστε να μην γίνονται πλέον διαβουλεύσει σε σκοτεινά δωμάτια. Εγώ και το δικό μου το κόμμα, η δική μου πολιτική ομάδα θα αγωνιστούμε για μια Ευρώπη που θα ανήκει στου ανθρώπου. Για εμά, για του χριστιανοδημοκράτε, σήμερα είναι η μέρα μια νέα αρχή. Τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε, τώρα θέλουμε ένα νέο μέλλον με την Ursula von der Leyen ω πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε Βέμπερτ. Η πρόεδρο ε, Γκαρσία πέρε Ιράτσε ε, από του τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φοντερ Λάγεν. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, μια ιστορική ημέρα. Κρατάμε στα χέρια μας το μέλλον της Ευρώπης. Η πολιτική μου ομάδα, η οποία ε, εξ αρχής ε, ήταν φιλοευρωπαϊκή και έχει στο DNA του ε, το ευρωπαϊκό ιδεώδες ε, αισθάνεται ε, υπεύθυνο, ε, αισθάνεται υπευθυνότητα και απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα θέσουμε τις βάσεις για ένα μέλλον βιώσιμο για όλους τους Ευρωπαίους και όλες τις Ευρωπαίες. Επιτρέψτε μου να θυμηθώ σήμερα έναν μεγάλο Ευρωπαϊστή που πριν από 40 χρόνια πήρε το λόγο σε αυτό το κοινοβούλιο, ο Μπίλι Μπραντ μετά τις ε, ε, πρώτες ε, άμεσες εκλογές ε, μίλησε για κάτι που σήμερα πρέπει να υπεθυμίσουμε. Έλεγε ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία προχωράει με πολύ αργό ρυθμό ε, και ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν άμεσες ε, εκλογές. Αυτό ήταν καλό, αλλά παρόλα αυτά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνονταν να είναι πολύ μακριά από τους πολίτες και έλεγε πρέπει να δουλέψουμε πέρα από γεωγραφικές και ιδεολογικές διαφορές, να δουλέψουμε έτσι ώστε να λύσουμε τα προβλήματα και κυρίως για να μπορέσουμε να ε, συνδεθούμε με τους νέους. 40 χρόνια μετά ε, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ αυτή η συζήτηση. Αυτά τα λόγια είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Δυστυχώ με πολύ αργό προχωράει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Είχαμε πολλές αυταπάτες από ό,τι φαίνεται. Ε, είχαμε βάλει πολλές ελπίδες στη διαδικασία Spitzenkandidat. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία δεν μπορεί να οπισθοδρομήσει. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, ακούμε προσεκτικά την δέσμευσή σας κυρία Φόντερ Λάγεν σχετικά με την αναβίωση της σωστή της διαδικασίας Spitzenkandidat. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και αυτό πρέπει να, γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι πριν σας δώσουμε το αξίωμα της Προέδρου. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε μπορέσετε να ηγηθείτε αυτής της αλλαγής που μας ζητούν οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι νέοι. Ε, θέλουμε ε, έναν χάρτη ο οποίος να δείχνει τις πραγματικές προθέσεις, ε, την πραγματική βούληση για να προχωρήσουμε. Θα πρέπει η κλιματική αλλαγή να μας απασχολήσει και μάλιστα να νομοθετήσουμε. Είναι απαραίτητη νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει οπωσδήποτε να αναλυφθούν δεσμεύσεις όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών. Χρειάζεται διαφάνεια για όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε ε, που δέχεστε την δημιουργία ε, ταμείου για την ορθή μετάβαση. Επίσης ε, χαιρόμαστε που μιλάτε για την βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας αυτή θα πρέπει να προέρχεται από δημόσιου πόρους. Όταν συζητάμε και όταν συζητούμε τα θέματα ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο εξάμεινο, ε, ε, οπωσδήποτε θέλουμε κάτι παραπάνω. Δεν θέλουμε να κυρώνονται για υπερβολικό έλλειμμα κυβερνήσεις οι οποίες προσπαθούν να κάνουν πολιτικές οι οποίες προστρέχουν στις ανάγκες του κόσμου, που βοηθούν τους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν Χαιρόμαστε γιατί μιλάτε ε, στις προτάσεις σας για ευελιξία όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές. Τέλος, πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε που αναφέρεστε στην υποστήριξη του κοινωνικού πυλώνα και αναφέρεστε επίσης στην εγγύηση για τους νέους και για τα παιδιά. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε κυρία Φοντερ να αγωνιστούμε περισσότερο ενάντια στην φτώχεια. Ο καθένας από το μετερίζει του, ο καθένας από αυτό που μπορεί να κάνει. Εσείς ε, θέλετε οι φόροι να συμβάλλουν από ό,τι μας είπατε σε αυτή τη διαδικασία αλλά έχετε σκεφτεί κάποιο συγκεκριμένο ποσό ε, με ποιο τρόπο θα προστατέψουμε τους εργαζόμενους κυρίως αυτούς που εργάζονται στις νέες πλατφόρμες χρειάζεται νομοθέτηση όσον αφορά τα θέματα αυτά επίσης όσον αφορά την αναφορά σας στην ισότητα των φύλων είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος η πολιτική μου ομάδα έχει συγκεκριμένη πολιτική να ε, ε, υπάρξει συγκεκριμένη λοιπόν στρατηγική για την ισότητα των φύλων και οπωσδήποτε αυτό που είπατε για τη σύνθεση του ε, Κολεγίου των Επιτρόπων είναι οπωσδήποτε μια καλή αρχή. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός που να διασφαλίσει αυτήν την λειτουργία. Πιστεύω ότι θα μας καθησύχαζε πολλές και πολλούς εδώ στην αίθουσα εάν μας ε, ε, λέγατε ότι ε, θα, όσον αφορά το κράτος δικαίου, ότι θα συνεχίσετε την πορεία που ξεκίνησε ο Φραν Τίμερμαντ όσον αφορά το κράτος δικαίου. Πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε για αλληλεγγύη, πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε ε, για αυτές ε, τις ανθρωπιστικές ε, λεωφόρους και διάβλους όσον αφορά τη μετανάστευση. Αλλά κυρίως πρέπει και πρωτίστως να σώσουμε την ζωή των ανθρώπων. Θα πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα διάσωσης που να μην κυρώνει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δεν είναι δυνατόν Λοιπόν να δεχτούμε μια ε, ε, θεσμική κρίση η οποία θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Αλλά θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον, αλλά με ασφάλεια, με τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Η ομάδα μου θα πάρει μια απόφαση το απόγευμα με την ελπίδα ότι άνδρες και γυναίκες θα έχουμε το κοινό όραμα ε, και είμαι βεβαία ότι θα συναντηθούμε σε αυτήν την διαδρομή οικοδόμησης, σε αυτό το τόσο σημαντικό όραμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Τσιόλος, έχετε το λόγο. Κυρία υποψήφια πρόεδρε, το Κοινοβούλιο ε, δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικό και τόσο εμπλεκόμενο, γνωρίζοντας τις ευθύνες και έτοιμο να τις αναλάβει πλήρως. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Συμβούλιο το οποίο σας ανέδειξε είναι ένα διχασμένο Συμβούλιο. Ε, συνήθει μετά από ένα πακέτο για να εξασφαλίσει ένα συμβιβασμό μετά από μακρέ διαπραγματεύσει. Και λυπούμε που η ισορροπία ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντανακλάται σε αυτό το πακέτο και ελπίζω ότι θα ε, αποκατασταθεί όταν ανατεθούν τα χαρτοφυλάκια στο Σώμα των Επιτρόπων. Σήμερα εδώ δεν υπάρχει κανένα πακέτο. Υπάρχει μία ε, υποψηφιότητα, η δική σα, με βάση τι δεσμεύσει που τις έχουμε ενώπιόν μας. Σήμερα ε, ε, αναζητείται μια πλειοψηφία που να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να προχωρήσει και να ανταποκριθεί στις ε, απαιτήσει που αναφέρθηκαν. Η ιδέα του Spitzenkandidat, δηλαδή της ε, ε, εκλογής μέσα από την εκλογή όλων των πολιτών, δεν οδηγήθηκε, ε, δεν τερματίστηκε. Αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει στο τέλος να πετύχει και χαίρομαι που αναλάβατε την ιδέα ενός, μιας διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που να οδηγήσει σε πέρα σε αυτή την εκδημοκρατικοποίηση. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η διαπραγμάτευση μαζί σας από τις Ευρωπαϊκέ ομάδε ήταν με βάση μια κοινή πολιτική πλατφόρμα αυτών των ομάδων. Εάν εκλεγείτε, αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να μα προσφέρει ένα πλαίσιο εργασία που να είναι κοινό και διαφανέ, ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ε, ε, στόχου σαφείς για την επόμενη πενταετία. Η ομάδα μα είναι έτοιμη να σα υποστηρίξει στο μέτρο στο οποίο θα αναλάβετε την ανεξαρτησία και την ε, δύναμη πρόταση για την ανανέωση της Ευρώπης οι ε, δεσμεύσεις που αναλαμβάνεται σήμερα αν είναι πιο σαφείς και πιο προευρωπαϊκές τόσο πιο πολύ θα είμαστε σε θέση να κτίσουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες μια Ευρώπη που να ε, ξαναδώσει ε, την ελπίδα και την αυτοπεποίθηση. Στις ε, εκλογέ υπήρχε ένα πνεύμα κατά ε, αντιευρωπαϊκό και θα έθετε την Ευρώπη σε δυσκολίες. Αυτό το τσουνάμι όμως δεν έγινε ε, και οι προευρωπαϊκές δυνάμεις είναι δυνατές σε αυτό το νέο σώμα. Δεν πρέπει όμως να απογοητεύουμε τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που είπαν ναι σε αυτή την Ευρώπη. Αυτοί αναμένουν ότι αυτή θα προασπίσει το κράτος δικαίου χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε τα εκατομμύρια των νέων που ήρθαν να ψηφίσουν και έστειλαν μια έκκληση για την καταπόλεμηση της αλλαγής του κλίματος. Δεν πρέπει να απογοητεύσουμε τα εκατομμύρια των επιχειρήσεων, των μισθωτών και των γεωργών που αναμένουν έτσι ώστε η Ευρώπη να γίνει μια πραγματική ευκαιρία σε έναν ανοιχτό κόσμο. Μια Ευρώπη που να κτίσει μια ε, οικονομία προς τους πολίτες για να ενσωματώσει την οικολογία, την κλιματική ισορροπία, την αηφορία αλλά και τις νέες τεχνολογίες τεχνολογίε για την ψηφιακή στατική ως ευκαιρίες και όχι προκλήσεις και περιορισμούς. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να βγει από τους αριθμούς και από τη γραφειοκρατία και να δημιουργήσει ευημερία για τον κόσμο. Ωστόσο, πάνω απ' όλα, αναμένουμε από εσά, κυρία Ορσολαβαντελάιν, μια καθοδήγηση ευρωπαϊκή, προευρωπαϊκή πραγματικά. Η Ευρώπη δεν είναι απλά διοίκηση, είναι πάνω απ' όλα μια πολιτική φιλοδοξία των πολιτών. Εάν ε, θα ε, σας ψηφίσει αυτό το σώμα το οποίο ε, σας εύχομαι, θα, είμαστε, θα θέλουμε να ακούσουμε επιχειρήματα που να σας πείθουν ότι πολλές αλλαγές δεν, θα ακούσετε ότι δεν θα γίνονται, αλλά εσείς θα πρέπει να τις καταστήσετε δυνατές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάμπερτ, έχετε το λόγο. Καίγεται το κοινό μας σπίτι. Καίγεται ε, από την ε, βιοπικιλότητα που χάνεται, από τις, ε, τους φυσικούς πόρους που εξαντλούνται, από την ολοένα και αυξανόμενη φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση απέναντι σε αυτήν την επίγουσα κατάσταση η καλή θέληση και οι καλές προθέσεις γενικής φύσεως δεν αρκούν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε πορεία, έστω και αν πρέπει να ε, έχουμε κατά μέτωπο αντίθεση με αυτούς που ε, αντιστέκονται. Τον Μάιο εξελέγει ένα νέο κοινοβούλιο και σήμερα βρισκόμαστε απέναντί σας κυρία Φόντερ Πριν από τρεις εβδομάδες ούτε καν ξέρατε ότι θα είσαστε ε, υποψήφια ε, για αυτήν την τόσο σημαντική θέση, πρώτη ε, θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο αναγκαστήκατε να σκεφτείτε κάποια πράγματα και επομένως θεωρούμε θεωρούμε ότι αυτά που μας είπατε σήμερα και τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν τα λεγόμενά σας ε, ε, αποτελούν πραγματικά μια πολύ καλή πρόοδο. Ε, χαιρόμαστε για αυτά που είπατε όσον αφορά την ισότητα ανδρών γυναικών. Επίσης το γεγονός ότι αναφέρεστε στην μείωση των εκπομπών μέχρι το 2050 καθώς επίσης και αυτή είναι την φορολόγηση των εκπομπών που αποτελούσε μέχρι τώρα ταμπού για την πολιτική οικογένεια από την οποία να προέρχεστε. Αλλά θα ήθελα να σας πω το εξή. Γιατί ας πούμε η ε, κλιματική στόχη απέναντι σε μια τόσο κατεπίγουσα κατάσταση ε, ε, προτείνεται δύο φάσεις και όχι άμεση αντιμετώπιση. Επίσης, γιατί αναφέρεστε στην αιρεσιμότητα. Υπογραμμίζεται ορθώς ότι σε αυτήν την κλιματική μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και θα πληγούν από μια ε, μη αντιμετωπιστήσα ε, κατάσταση. Ε, επίσης θα πρέπει και η φορολόγηση να γίνει πραγματικά δίκαιη το πρόβλημα δεν είναι μονάχα βεβαίω το κλίμα. Ας ε, μιλήσουμε για την ε, ε, βιοπικιλότητα. Κατά την έννοια αυτή, η κοινή γεωργική πολιτική που παίρνει τα περισσότερα χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει καταστροφική επίπτωση και ε, καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα βρει μεγάλη αντίσταση από αυτούς που αποφελούνται από το σύστημα. Ε, επίσης, ε, η εμπορική πολιτική λέτε ότι σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ρήτρε για την βιώσιμη ανάπτυξη. Από την άλλη μεριά βέβαια αυτές οι ρήτρε υπάρχουν ήδη και από την άλλη πλευρά εσείς εσείς ε, ε, κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά δικαιώματα των επενδυτών. Ε, επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι απαράδεκτο να βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολοκληρωτικά καθεστώτα ή σε καταλημμένα κράτη έτσι ώστε να κάνει αυτήν την πολιτική. Αυτές οι συμφωνίες δήθεν με την ακτοφυλακή της Λιβύης δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. Αυτή η συμφωνία που λέτε κυρία Φόντερ Λάγεν ε, υπάρχει ήδη ε, και επομένω. μην κομίζετε γλάφκα στις Αθήνα. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν ήδη και τα στοιχεία αυτά και τα θέματα αυτά έχουν υπερψηφιστεί εδώ στο Κοινοβούλιο και με μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα. Όλα αυτά που λέτε παραμένουν ασαφή. Το ζήτημα είναι να αλλάξει πραγματικά η παρτίδα. Το ζήτημα είναι να δώσουμε την δυνατότητα ε, αυτοί, αυτές οι ε, χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Πολωνία που καταπατούν διαρκώς το διαχωρισμό των εξουσιών να μπουν στη θέση τους. Ε, επομένως, ε, ε, κατεπίγουσα κατάσταση όσον αφορά τα πολιτικά, τα, κοινωνικά, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή οι οικολόγοι και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που είπαμε, δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε να κυβερνείτε, το τιμόνι για να κυβερνήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ, ξέρετε, κυρία Βοντερλάγεν ότι έχουμε μια φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία. Ωστόσο, δεν έχουμε χρόνο ακόμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτές τις συμμαχίες. Και επίσης δεν ακούσαμε από τη μεριά σας ε, την ε, πραγματική βούληση για μια τέτοια ε, συμμαχία. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι κλείνετε το μάτι και προς εθνικιστικές, λαϊκιστικές ας πούμε αρχές. Εάν εκλεγείτε σήμερα, σας διαβεβαιώ ότι θα είμαστε από απολύτως ανοιχτή να μας πείσετε ε, ε, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι και σε δημοκρατικό και σε κοινωνικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο οι προτάσεις σας ε, θα είναι σωστές. Δηλαδή σωστές σε κάθε επίπεδο από αυτά που χρειάζεται η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μόιτεν έχει το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κυρία Φοντελάν. Σήμερα σε αυτή την αίθουσα έχουμε να λάβουμε μια πολύ σημαντική απόφαση. Πρόκειται για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα αξίωμα που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Για το αξίωμα αυτό ε, είναι κατάλληλο μόνο κάποιο που έχει όλα τα προσόντα. Κυρία Υπουργέ, με κάθε σεβασμό προ το πρόσωπό σα, εμεί από την πολιτική ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, μετά από ενδελεχή εξέταση του όλου θέματο, καταλήξαμε στο ότι εσεί δεν είσαστε κατάλληλοι για το αξίωμα αυτό. Και θα το εξηγήσω. Καταρχήν, εμεί, οι Γερμανοί, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε διάφορα θέματα, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε την εμπειρία μας. Ήσασταν υπουργό Οικογένεια, ήσασταν υπουργό Κοινωνικών Θεμάτων και τέλος ήσασταν υπουργό Άμυνα στη Γερμανία. Σε κανένα από αυτά τα αξιώματα δεν υπηρετήσατε ικανοποιητικά το λαό, του πολίτε. Δεν θέλω τώρα να σα πω ακριβώ που αποτύχατε, αλλά ξέρετε τι κάνατε. Κάνατε στρατηγικές οικονομίε στο στρατό, το γερμανικό, που σήμερα αυτός ο στρατός δεν είναι σωστά εξοπλισμένος και δεν μπορεί να επερασπιστεί τη χώρα. Και γι' αυτό το λόγο, εάν εκλεγείτε, ε, είπατε ότι θα παραιτηθείτε από Υπουργό Άμυνα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οι γερμανικές κυβερνήσεις κατά το παρελθόν είχαν διάφορου ε, πολιτικού ε, που του έστειλαν σε θέσει στι Βρυξέλλες. Σήμερα όμω αυτό πια δεν μπορεί να ισχύει Κατά την δική μας άποψη δεν υπάρχει τίποτα που να μας πείτε ότι θα κάνατε καλύτερη δουλειά στη θέση του πρώτου Επιτροπής από ό,τι κάνατε στα παλαιότερα αξιώματά σας. Όλα αυτά τα νεφελώδη που υποσχεθήκατε, το Α, το Β και πολλές φορές όλες οι αντιφάσεις στις οποίες υποπέσατε, όλα αυτά οδηγούν στο να μην είμαστε μόνο εμείς επιφυλακτικοί απέναντί σας. Οι ε, αριστεροί και οι ε, φιλελεύθεροι αναφέρονται στο άρθρο στο ECR επίσης έχουν επιφυλάξεις ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τους μετανάστες. Αντιφάσεις λοιπόν. Και σήμερα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι μας είπατε πολλά ευχάριστα, ο καθένας να ικανοποιηθεί, ο καθένας να ακούσει αυτά που θέλει. Σήμερα λοιπόν, ε, αλλά και όλες αυτές τις ημέρες ε, που προσπαθείτε να μας πείσετε, δείχνετε μια πολιτικό που θέλει να ικανοποιεί όλους. Ο Τζάκελ και ο Χάιντ είσαστε τελικά και προσπαθείτε με τον τρόπο αυτό να συγκεντρώσετε ψήφους. Το πρόβλημά σας με όλα αυτά είναι ότι δυστυχώς δεν είσαστε πιστικοί, δεν έχετε το όραμα ενός σύγχρονου ανθρώπου που πραγματικά να υπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ένωση που να εκπροσωπεί τα κράτη της. Του αντίον, εσείς τι κάνετε, υπόσχεστε ακόμα μεγαλύτερη συγκεντρωτική μορφή, ακόμα περισσότερους φόρους και ε, με τον τρόπο αυτό ε, δυστυχώς υποπίπτεται σε αντιφάσεις ε, και από ό,τι φαίνεται όμως δυστυχώς δεν το συνειδητοποιείτε. την προηγούμενη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων σας έκανα κάποιες ερωτήσεις και εσείς δύο ερωτήσεις δικές μου ούτε καν τις απαντήσατε και την τρίτη που απαντήσατε εκεί ήσασταν παντελώς μη ικανοποιητικοί. γι' αυτό λοιπόν αυτά που μας είπατε σήμερα που είναι και σοσιαλιστικά πρέπει να πω εμάς δεν μας πείτε. και για το λόγο αυτό εμείς θα σας καταψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Φίτο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, κυρία Βαντερλάγεν, ε, και με μεγάλη προσοχή σας είχα ακούσει όταν ήρθατε και στην ε, συνεδρίαση της ομάδας μας. Στη σημερινή, μας, στη σημερινή σας ε, παρέμβαση οι θέσεις σας έχουν αρκετά τροποποιηθεί σε σχέση με αυτά που μας είπατε την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ θα ξεκινήσω